Και άκουσα και τον κύριο Μιλάνα, έφυγε τώρα, αλλά αναφέρθηκε στην ιδετοκαλλιέργεια και το επέλεγαν αυτά και άλλοι συνάδελφοι, ο την Αντινόρο και άλλοι. Νομίζω ότι θα πρέπει να το τονίσουμε. Η Κάρμεν μίλησε για τη θαλάσσια πολιτική και έχει δίκιο, εξηγώντα ότι δεν είναι μόνο η δική μας επιτροπή η οποία είναι αρμόδια και καλείται εδώ, αλλά και η επιτροπή η η επιτροπή για τις μεταφορές. Υπάρχουν πολλές επιτροπές που είναι αρμόδιες για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και αυτό είπε και ο κ. Στορκάς και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε. Τώρα για τις προσωρινές παύσεις, ε, συμφωνώ με την κυρία Φράγκα, η οποία προτείνει την διατήρηση αυτών των προσωρινών παύσεων, των προσωρινών παροπλισμών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ε, ενισχύσεις και τις σχετικές διακρίσεις, ε, γιατί να θέσουμε τώρα το κατόφλι στους 100.000 κατοίκους, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Κατά την ε, άποψή μου δεν έχει κανένα νόημα, δεν είναι ένα κριτήριο που μπορούμε να το δεκτούμε αυτό. Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση στην αποθεματοποίηση, το είπα αυτό στην αρχή, είμαι υπέρ της ενίσχυσης στην αποθεματοποίηση και ενίσχυση. Ε, ναι, αυτό είναι κρίκος της αλυσίδας, Τον να ενισχύσουμε το ρόλο τη μεταπητική βιομηχανία. Ε, δεν έχουμε μόνο στην Ισπανία τη βιομηχανία, αλλά και σε άλλε χώρε και νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό, γιατί αυτό ο κρίκο αλυσίδα είναι σημαντικότατο. Και επίση έχουμε και το άρθρο 71, πρέπει να επιμείνουμε εκεί, στη θέση τη εμπορία, στη θέση εμπορία, με συγχωρείτε, και στην καινοτομία. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Θέλω να έχουμε πολύ συγκεκριμένες ε, δράσεις. Συμφωνώ λοιπόν μαζί σου κύριε Ρόντουστ. Ε, υπογράμμισες ε, το ενδιαφέρον των συμπράξεων, τη συνεργασία των αλλιών με τους επιστήμονες. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό. Επίσης, αναφέρθηκες στους εμπειρογνώμονες. Εγώ δεν έχω και τόση εμπιστοσύνη στους εμπειρογνώμονες επί της αρχής. Γιατί, εντάξει, μπορεί να έχουν γνώσεις, αλλά εγώ κάποια δυσπιστία. Ναι, εμπειρογνώμονε, ναι, μένα, αλλά υπάρχει και πραγματικότητα επιτόπου. Σε ό,τι αφορά τον εξυγχρονισμό του στόλου, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και όπω και να έχει, δεν ε, μιλάμε εδώ φυσικά για αύξηση τη αλεία. Ε, ε, των αλλιευμάτων πρέπει να διατηρήσουμε τα παθήματα και να προσέχουμε την βιοπικιλότητα και το περιβάλλον. Και μια άλλη ενδιαφέρουσα παρατήρηση που υποθήκε από το Στρούαν. Συμφωνώ απόλυτα για τον να μια καταγραφή της πλεονάζουσας ε, ικανότητας. Όμως η Ευρώπη είναι μεγάλη και υπάρχουν ε, κάποια μέρη στα οποία βλέπουμε ότι υπάρχει τέτοια πλεονάζουσα ικανότητα, αλλά δεν ισχύει παντού. Γι' αυτό είμαστε υπέρ της περιφερειοποίησης και θέλουμε να ακολουθήσουμε και αυτή την προσέγγιση στην περιφερειοποίηση. Τώρα, πρόεδρε, τέθηκε ένα ουσιαστικό πρόβλημα, η διαφορά μεταξύ των διάφορων θαλάσσιων περιοχών και των ε, αλλιευμάτων, ε, γιατί είναι διαφορετικό να έχουμε μια πολιτική που θα καλύπτει ε, όλη την επικράτη από τη Βαλτική στη Μεσόγειο, δεν έχουμε παντού τέτοια προβλήματα και έχουμε και τον αυξηνό πόντο, έτσι. Πρέπει να διαφοροποιήσουμε λοιπόν. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να διαφοροποιήσουμε το πρόβλημα αυτό, κυρίω ό,τι αφορά στο θέμα τη πλειονότητα ικανότητα, αλλά και σε άλλου τομεί. Ε, γι' αυτό είναι ενδιαφέρουσα η περιφερειοποίηση. Euh, Για την ανανέωση του στόλου, επανέρχομαι. Σα υπενθυμίζω ότι πραγματικά όπως και εμείς ηλικιώνεται. Και ο ευρωπαϊκός στόλος σε 10 χρόνια θα είναι 10 χρόνια γυρεότερος. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να έχουμε κατά νου και αυτό το πρόβλημα. Θέλουμε να διατηρήσουμε την παράκτη αλία, την αστεχνική αλία. Θέλουμε να τη διατηρήσουμε στο μοντέλο αλίας μας ή όχι. Αυτή είναι η φιλοσοφία της μεταρρύθμισης για τη βοήθεια στην αποδοματοποίηση Σας ε, το είπα, είναι υπέρ. Στην Εθνική τον αναφέρθηκε σε πολλά πράγματα. Είπε ότι δεν ε, ήταν υπέρ ε, στο να έχουμε υποχρεωτικέ μεταβιβάσει με ελευτικές παραχωρήσεις, ε, αλλά από ό,τι είπατε θέλετε ε, θελούσιες, αν κατάλαβα καλά αγαπητέ συνάδελφοι. Επίση, είπατε ότι είσαστε υπέρ η μείωση των απορρίψεων να είναι προοδευτική και να συνοδεύεται από ενίσχυση, αν κατάλαβα καλά, για να φτάσουμε σιγά σιγά σε αυτό το στόχο γιατί φυσικά όλοι θέλουμε να φτάσουμε στην μηδέν απορρίψεις, όλοι συμφωνούμε. Αλλά δεν θα μπορέσουμε να το πράξουμε παρά σταδιακά, μέσω της επιλεκτικότητας και δημιουργώντας υποδομές που σε επιτρέψουν κάτι τέτοιο, κάτι που δεν υπάρχει σήμερα. Λοιπόν, ο κύριος Νάρα Γκορμπάστικ φαίνεται ότι συμφωνεί μαζί μου για την υποστήριξη στην ανανέωση των κινητήρων. Λυπάμαι, αλλά εγώ ερμηνεύω την ε, πρόταση της Κομισιόν ε, ως ε, περισσότερο μία ενίσχυση στη μετατροπή παρά στην αλία. Έτσι είναι, με συγχωρείτε, λόγω της το ερμηνεύω. Και ο κύριος και επέμεινε επίση στην αναγκαιότητα εξυγχρονισμού των σκαφών για να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια για τους ναυτικού. Γιατί είναι πολύ δύσκολο επάγγελμα το επάγγελμα του ναυτικού. Δηλαδή δεν μιλάμε πάλι εδώ για να έχουμε περισσότερη αλίευση, αλλά να αλίευουμε καλύτερα, με πιο ευφυή τρόπο. Σήμερα αλίευουμε πολύ, αλλά δεν είναι άπειροι οι πόροι. Ο κ. Κούν είπε ότι θέλει αυτά τα κονδύλια να καλύπτουν και την ανταγωνιστικότητα του τομέα. Ναι, είναι λογικό, σταθεροποιώντα ε, την αλία, νομίζω ότι έχετε δίκιο, αλλά ήσασταν υπέρ και του εξυγχρονισμού, κατάλαβα καλά. Και αυτό εγώ θα το αποκαλούσα F.E. E, ανανέωση. Και επίσης έχουμε και ανάπτυξη και της καλλιέργειας. Ο κύριος Αντινόρο δήλωσε την, εκ νέου την υποστήριξή του στην υδατοκαλλιέργεια, ε, θα επιμείνουμε σε αυτό. Και ο κύριος ε, Γκάλαγκερ. Σε αυτά που είπε, νομίζω ότι είναι καλύτερη η αλήθεια σήμερα, συμφωνώ. Αλλά πιστεύω επίση να είμαι κάπως, ανώ, κάπως ε, αγαθός αλλά πιστεύω ότι κάπως σε στο μίσο, όπως στη Γεωργία Ήδη Οι διαλύσεις έχουν συνειδητοποιήσει ότι είναι αναγκαίο σήμερα παρά ποτέ πολύ περισσότερο σήμερα παρά ποτέ να σεβαστούν τους κανόνες. Οι αλήθεια είναι ήδη υπεύθυνοι, αν και μερικές φορές ε, ξέρουμε ότι οι ενισχύσεις ευνοούν ε, Ευρωπαίους αλείς, ε, και μερικές φορές δεν σέβονται τους κανόνες, όμως νομίζω ότι τώρα είναι στη διαδικασία συνειδητοποίηση πως αν συνεχίζουν να παραβιάζουν τους κανόνες, ε, ε, τότε ουσιαστικά σκάβουν το λάκκο τους. Έχουν αρχίσει λοιπόν να εξελίσσονται προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτά ήθελα να απαντήσω στους αδέλφους Κύριε Τοκάρσκι, μπράβο για το εγχείρημα να μας πείσετε, λυπάμαι όμως, αλλά εγώ δεν πείστε από επιχειρηματά σας. Σας το επαναλαμβάνω. Για μένα ουσιαστικά το Ταμείο παρουσιάζεται ως μία ενίσχυση στη μετατροπή και όχι ενίσχυση στην αλία. Σε ό,τι αφορά τώρα την έκθεση του λεκτικού συνεδρίου. Το αναφέρα και χτες, ε, τώρα η έκθεση του λεκτικού συνεδρίου, είτε στην Γαλλία είτε στις Βρυξέλλες, είτε κάπου αλλού. Με πολλού τρόπου μπορούμε να την ερμηνεύσουμε. Δεν έχουμε απριόρι, την ερμηνεύουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Πρέπει κάποιο λοιπόν να ξέρει να διαβάσει την έκθεση αυτή. Έχουμε κάποιε αιτιολογημένε συστάσει, αλλά αν διαβάσουμε δύο εκθέσει, ε, τι εκθέσει μάλλον το ένα δίπλα στον άλλο, δεν θα έχουμε την ίδια ανάλυση, σα διαβεβαιώ. Σα ευχαριστώ λοιπόν για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων, αγαπητοί συνάδελφοι, και φυσικά περιμένω και τι γραπτέ σα συνεισφορέ αλλά να επαναλάβω αυτό θα γίνει ανάλογα με την πρόοδο που θα σημειωθεί και στο, στο βασικό κανονισμό αλλά και στον κανονισμό για την ΚΟΑ. Γιατί θα πρέπει να εργαστούμε παράλληλα σε αυτές τις εκθέσεις. Μάλιστα. Είμαστε στο σημείο 13, αλλά να σας πω ότι έχουμε μία ώρα και δέκα λεπτά για τρία θέματα. Εδώ βρισκόμαστε για να συζητάμε, αλλά Κοιτάξτε, όταν ε, αρχίζουμε ένα σημείο της ημερησίας διάταξης και μόνο ένας, δύο, τρεις ε, ζητούν το λόγο, εγώ του αφήνω περισσότερο χρόνο γιατί υπολογίζω το χρόνο που θα χρειαστούμε. Αν Όμω όσο συνεχίζεται η συζήτηση ζητούν 10-11 άτομα το λόγο, είναι αδύνατο ο καθένα, ε, όπω συνέβη στο προηγούμενο σημείο να μιλάει 7-8 λεπτά γιατί θα φτάσουμε στα 80 λεπτά δεν είναι δυνατόν. Δύο προτάσει. δύο παρακλήσεις αν θέλετε. Ο καθώς ε, προχωράς τη συζήτηση, εντάξει μπορεί κάποιο να σκεφτεί ότι θέλει το λόγο, αλλά αν ζητήσετε το λόγο στη μέση της συζήτηση, μιλήστε μισό λεπτό. Αλλιώ ζητήστε το λόγο από την αρχή για να μπορέσω και εγώ να δω πόσο χρόνο θα δώσω. Και δεύτερον, ε, από τη στιγμή που δεν μπορούμε να έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μα, ε, να περιοριστούμε στα 2-2,5 λεπτά και θα πρέπει δυστυχώ να σα πω να ολοκληρώσετε, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να εργαστούμε αλλιώ, αλλά για το μέλλον να προσπαθήσετε σας παρακαλώ να ζητάτε το λόγο. Στο προηγούμενο σημείο ζήτησαν τρει, μίλησαν έντεκα. Πώ να υπολογίσω εγώ το χρόνο, είναι αδύνατον. Λοιπόν, Σήμερα 13 ορισμένα μέτρα και των χωρών πίσω επιτρέπουν τη εξαγωγή μη βιώσιμη αλληλεία με στόχο τη διατήρηση των αποθεμάτων χθείων. Ο κύριος ε, Γκάλεκερ είναι ορμόδιο συζητητής. Είχαμε μία πρώτη τελεγή απόψη. Αν έχετε το λόγο να μας παρουσιάσετε το σχέδιο. Ε, thank you, President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζει η Επιτροπή την το απαγοητευτικό αποτέλεσμα μεταξύ παράκτιων ε, από τη συνεδρίαση του στο Ρέικεβικ των παράκτιων κρατών. Είχαν γίνει και άλλες συναντήσεις ε, και μετά υπάρχει κοινή δήλωση της Επιτρόπου Δαμανάκη και του Νορβηγού ε, Επιτρόπου Αλίας. Ε, το πρόβλημα δημιουργήθηκε μετά τις μονοπλευρές αποφάσεις Ισλανδίας και Φερών και τα παράκτια κράτη συναντήθηκαν 11 φορές χωρίς ε, ε, συμφωνία. Η Ισλανδία αύξησε το, ε, την αλία του σκουμπριού σε 156.800 το 2011, ενώ παλιά δεν είχαν σχεδόν καθόλου. Τα αλλιεύματα των φερών αυξήθηκαν σε 250.000 σε το 2011, από 25.000 είχαν 156 φορές αύξηση, δηλαδή σε δύο χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νορβηγία ε, ε συμμετείχαν επικοδομητικά στις ε, ε, διαπραγματεύσεις, όχι όμως η Ισλανδία και η Φερόες. Η αλία του σκουμπριού είναι πολύ σημαντική και για στο όλο πελαγίων ειδών, για τις παράκτης περιοχές, Βεβαίως τώρα η έλεγχη είναι πιο αυστηρή και υπάρχει συνεργασία και από τον κλάδο, ο οποίος καταλαβαίνει πολύ καλά ότι η βιώσιμη αλία είναι προς το καλύτερο συμφέρον τους. Απειλείται το συμφέρον τους όμως από τις δράσεις των άλλων χωρών, ε, των παρακτήων χωρών. Πιστεύω λοιπόν ότι η Κομισιόν δεν είχε εναλλακτική από το να θεσπίσει εμπορικά μέτρα για να δράσει προληπτικά απέναντι στις χώρες ε, που κάνουν ε, πρακτικές μη βιώσιμης αλίας. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Κομισιόν. Βέβαια δεν είναι αρκετά αυστηρή αν τη δούμε στις λεπτομέρειες. Αναφέρεται μόνο σε κυρώσεις σε σχέση με τα ψάρια που έχουν αληφθεί με τρόπους μη βιώσιμης αλίας. 4% έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε εκεί είναι σαν να μην κάνουμε τίποτα. Ε, ενώ η πρόταση της Κομισιόν περιορίζεται σε ό,τι αφορά τα ψάρια στόχος που τα ε, υπεραλλιεύονται και είχαμε μια συνάντηση για, με πρώτη ανταλλαγή ε, και είχαμε συνάντηση και με τους σκιώδεις και αποφασίσαμε να επεκτείνουμε το μέτρο πέρα από τα όρια της πρότασης της Κομισιόν. Θέλουμε να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής των μέτρων για τα ψάρια και τα λιευτικά προϊόντα ε, στη συνεδρίασή μας με τους Σκιώδης ακούσαμε καλές προτάσεις από την Κάρμεν Φράγκα, με την οποία είχα ζητήσει και από πριν, δεν μπορούσε να έρθει τότε, αλλά ε, έδωσε καλές προτάσεις και ε, επίσης η Ιζαμπέλα Λεβίν. Αυτά τα έλαβα πριν από τη συνάντηση σήμερα, τη συνεδρίαση σήμερα και η πρόθεσή μου είναι να τα συμπεριλάβω στην έκθεση. Εν ολίγης, κυρία Πρόεδρε, έχουμε εδώ μια σοβαρή κατάσταση να αντιμετωπίσουμε. Οι επιστήμονες λένε ότι η αλλιεύση 650.000 τόνων ε, επιτρέπει την ε, ανασύσταση αποθεμάτων. Τώρα όμως ε, η εκφόρτωση είναι ένα εκατομμύριο τόνοι. Τελείως ε, αδύνατον, δεν είναι βιώσιμο αυτό. Σε λίγα χρόνια δεν θα μπορούμε να ψαρεύουμε ε, στην περιοχή αυτή. Αλλά και αυτοί που κάνουν μη βιώσιμη αλεία και εκείνοι τα ίδια προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε. Πρέπει λοιπόν να δούμε και τις κυρώσεις υπό αυτό το πρίσμα Εδώ είναι ένα θέμα που αφορά όλη την Ευρώπη και τρίτε χώρες με τις οποίες έχουμε εταιρικέ συμφωνίες. Όλοι θα πληγούν, όλοι θα επηρεαστούν. Μακάρι να μην χρειαστούν τα αυστηρά μέτρα, αλλά θα πρέπει η Κομισιόν με την υποστήριξη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελπίζω, να είναι σε θέση να ενεργοποιήσει τα μέτρα όποτε χρειαστεί. Ελπίζουμε ότι θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα έτσι. Αυτά είναι κάποια σχόλια λοιπόν σε αυτό το στάδιο. Θα πρότεινα κύριε Πρόεδρε η νομική υπηρεσία να μας ενημερώσει γιατί ακόμα το εξετάζει, εξετάζει την πρόταση. Θα πάρουμε και τις άλλες τροπολογίες και μέχρι την Παρασκευή θα τις έχουμε όλες. Καλύτερα λοιπόν η προθεσμία κατάθεσης να παραταθεί μέχρι τη Δευτέρα για να προλάβουμε να εξετάσουμε τις τροπολογίες και να έχουμε και τη γνώμη της νομικής υπηρεσίας. Έχουμε χρόνο και παρόλα, παρόλη την παράταση θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε στη Σύνοδο του Μαρτίου. Ευχαριστώ κύριε Καλό και τέσσερα άτομα έχουν ζητήσει το λόγο. Λοιπόν, να κλείσουμε εδώ τον κατάλογο και σας παρακαλώ δύο λεπτά το πολύ. Κύριε Στίβενσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Γκάλαχερ παρουσίασε τη σοβαρότητα του προβλήματος. Εγώ κατανοώ την Κομισιόν γιατί οι νήσι Φερόες ήταν μέρος της Συμφωνίας των Παράκτιων Κρατών και παραβίασαν τη Συμφωνία οι Φερόες. Εμείς δεν μπορούμε όμως να εφαρμόσουμε κυρώσεις παρά μόνο για το συγκεκριμένο είδος, το οποίο είναι το σκουμπρί. Και εκεί, όπως είπε και ο κύριος Κάλαχερ, οι ε, εισαγωγές αυτού του είδους δεν είναι μεγάλες στην, ε, στην Ένωση, οπότε και οι κυρώσεις δεν θα έχουν νόημα. Όμως η Ισλανδία δεν ήταν ποτέ μέρος της Συμφωνίας Παρακτήων Κρατών, οπότε εκεί μπορούμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε όλα τα αλλιευτικά προϊόντα. Οριζόντια μέτρα Μπορεί να παραβιάζουμε τον ΠΟΕ, αλλά τουλάχιστον θα τους απειλήσουμε και θα δει και η νομική υπηρεσία αν μπορούμε να επεκτείνουμε τις κυρώσεις και πέρα από τα αλληλευτικά προϊόντα. Επίσης να εξετάσουμε επίσης πάλι το θέμα της προσχώρησης της Ισλανδίας στην Ένωση. Δεν μπορούμε εμείς να τους τρώνουμε το κόκκινο χαλί με συνοπτικές διαδικασίες για να μπουν στην Ένωση, ενώ αυτοί ε, κάνουν παράνομη άναρχη α, λαθρέα αλία. Αυτό είναι πειρατεία του χειρότερου είδους. Και υπάρχουν και συμφωνίες μεταξύ Κομισιών και Νορβηγίας, Φερόες και Ισλανδία και σε συνομιλίες και όλες απέτυχαν. Μετά από όλα αυτά θα πρότειναν η Επιτροπή να στείλει τον κύριο Γκάλαχαρ στην περιοχή, να πάει στο Ρεκιαβίκ και στις Φερόες να μιλήσει με τους Υπουργούς Αλίας και στις ε, δύο χώρες. Εγώ το έκανα όταν πρώτο ξεκίνησε το πρόβλημα, χωρίς αποτέλεσμα. Τώρα όμως που φτάσαμε σε αυτή τη θλιβερή κατάσταση, αν συμφωνεί και ο κύριος Γκάλαχαρ, θα ήταν πολύ καλό να το κάνει η Επιτροπή μας, να τον στείλει. Εξαρτάται από εσά και τους συντονιστές βέβαια να αποφασίσετε εάν κάτι τέτοιο είναι σκόπιμο. Ευχαριστώ, κυρία Φράγα. Θα είμαι σύντομη. Θέλω απλώ να ευχαριστήσω τον κύριο Γκάλακερ για τη διαθεσιμότητά του για να δούμε αυτό το θέμα ευρέω. Συμφωνώ απόλυτα με τι τροποπολογίε του. Ανεξάρτητα με το αν πρέπει και η νομική υπηρεσία να αναλύσει το νομικό σκέλο, αλλά κατανοώ ότι έχει διευρυνθεί το πεδίο δράση. Δεύτερον, σα ευχαριστώ προσωπικά που έχετε συμπεριλάβει σε δύο τροπολογίε τι δικέ μου προτάσει ε, να έχουμε διεύρυνση από διμερεί σε πολυμερή θέματα. Έτσι λοιπόν, ε, εγώ νομίζω ότι δύο τροπολογίες ε, που αφορούν τις περιφερειακές οργανώσεις αλίας είναι πολύ θετικέ και σας υποστηρίζω. Ευχαριστούμε κυρία Φράγκα και κυρία Λοβάν. Okay, I too would like... Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Ήταν πολύ καλή συνάντηση των σκιωδών. Υποστηρίζουμε επίσης την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής. Φυσικά θα ήθελα να γνωρίζω και τις νομικές συνέπειες αυτού, ότι δηλαδή θα πρέπει ίσως να προβλεφθεί η αμοιβαιότητα. Ε, ουδάλλως θα παραβιάσουμε τους κανόνες ΠΟΕ. Θέλουμε να παρατείνουμε και την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών μέχρι τη Δευτέρα ή και αργότερα, αν χρειάζεται αυτό διότι θέλουμε να πετύχει αυτό και όχι να αποτύχει. Ευχαριστούμε κυρία Ρόντος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ και η ομάδα μου θέλουμε να συγχαρούμε τον κύριο Γκάλαχερ και τους Σκιώδης επίσης. 11 φορές συναντήθηκαν χωρίς αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν τουλάχιστον εμείς Πολύ ε, πασχίσαμε για μία λύση, αυτό είναι σαφές. Έχουμε κανόνες στην Ένωση, αν δεν τηρούνται, τότε η άμυνα είναι οι κυρώσει και πρέπει να τις εφαρμόσουμε. Να συμφωνήσουμε με τον Πατ και να πούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε στα πλαίσια των κανόνων του ΠΟΕ. Θα τα δει αυτά η νομική υπηρεσία και θα μας πει, αλλά Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω ούτε χιλιοστό. από την Ευρωπαϊκή Ο κύριος Στουντίγιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά και που πέτυχε την ε, Γενική Συμφωνία αυτής της Επιτροπής, από όσο βλέπω. Κατανοώ ότι η έκθεση του κυρίου Γκάλακερ κατά κάποιο τρόπο εγκρίνει την πρόταση της Κομισιόν και όχι απλώς την εγκρίνει, αλλά προτείνει να πάμε και ακόμη παραπέρα. Πιστεύω ότι θα περιοριστώ στο να πω ότι η Κομισιόν ε, εξέτασε όλες τις νομικές πτυχές της πρότασης αυτής πριν από την προετοιμασία της και κατανοώ ότι η Κομισιόν πήγε όσο πιο μακριά μπορούσε σε σχέση με το τι μας επιτρέπει ο ΠΟΕ. Τώρα, νομίζω ότι κρεμεί η εξέταση της πρότασης από την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Θα περιμένουμε για να δούμε πώς θα δημορφωθεί τελικά αυτή η έκθεση και σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Γκάλακερ για να ολοκληρώσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την υποστήριξη που μου προσφέρουν. Ευελπιστούμε ότι μετά τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με αυτή την έκθεση, διότι είναι απολύτως αναγκαία. Ακούγοντας ε, τον, την Επίτροπο, και με όλο το σεβασμό που τρέφει για αυτήν, γιατί θέλω να ευχαριστήσω και την Επίτροπο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τις αρχικές ε, συζητήσεις ε, ανέλαβαν αυτή την πρωτοβουλία και χάρη σε αυτή την πρωτοβουλία τώρα εμείς μπορούμε να κάνουμε μια ισχυρή πολιτική δήλωση για αυτό το θέμα. Ως προς την υπόδειξη του Στρούαν Στίβενσεν γνωρίζετε Πρόεδρε ότι θα πάμε τις επόμενες εβδομάδες στην Ισλανδία και ε, ευελπιστούμε ότι θα συναντηθούμε με τον νέο Υπουργό Αλίας και πιστεύω ότι ήδη γνωρίζει τις ε, προτάσεις. Ε, φυσικά να συναντηθούμε και με εκπροσώπους των νήσων Φαρόε, αν αυτό χρειάζεται, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μια λογική ανταπόκριση. Την περασμένη εβδομάδα ε, ήμουνα σε μια διακοινοβουλευτική συνεδρίαση στην Νορβηγία και ζήτησα να συζητήσω με την Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων τελικά μπορούσα να δω τον Υπουργό Αλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων. Ανησυχούν πολύ διότι ε, πριν από δύο χρόνια ε, καταργήθηκαν και αυτές οι περιορισμένες κυρώσεις, δηλαδή δεν άφηναν, δεν επέτρεπαν την εκφόρτωση των σκαφών που αλίευαν κοντά στην Νορβηγία. Πολύ βασικό θέμα, διότι όταν εκφορτώνται τα αλίευματα, ε, καταψύχονται και μεταποιούνται από την τοπική βιομηχανία Και τώρα ε, σίγουρα θα περιμένουν με αγωνία την έκβαση των συζητήσεων για αυτήν την έκθεση, διότι τους απασχολεί αυτό το θέμα. Ε, ε, σχετικά με τις τροπολογίες, είπατε για τη Δευτέρα, νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε την ημερομηνία του Μαρτίου. Όλοι γνωρίζουν για ποιου λόγους. Ας δούμε τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο με τις τροπολογίες και βλέπουμε. Ευχαριστούμε κύριε Καλακέρα. Βέβαια, θα έχουμε μεγαλύτερη προθεσμία για την Δευτέρα 5 του μηνό στις 12 το μεσημέρι. Όχι στις 2 του μηνό, στις 5 του μηνό. Διευρύναμε την προθεσμία λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το επόμενο σημείο είναι το σημείο 14. Ο κύριο Φεραίρα δεν έχει φτάσει ακόμη και μας ζήτησε να δούμε το τελευταίο σημείο, το σημείο 15 της κυρίας ε, Λοβέν ε, συμφωνεί και μάλιστα βρίσκεται και εδώ και ο αρμοδίο του Περσίστη. Λοιπόν, να περάσουμε στο σημείο 15, εξωτερική διάσταση τη κοινή ελευτική Και Έχουμε μια προσκεκλημένη παρουσίαση συγκήτρια στις 24 Ιανουαρίου των Γραφοργασίας και θα ακούσουμε μια παρουσίαση της κυρία Μουτανέτ, η οποία είναι συντονίστρια της Μαυριτανίας 2000, ε, οργάνωση που εκπροσωπεί γυναίκες που εργάζονται στη μεταπιτική βιομηχανία αλευτικών προϊόντων στη Μαυριτανία. Και χωρίς χρονοτριβή να δώσουμε καταρχήν το λόγο στην κυρία Λοβέν και κατόπιν την κυρία Μουκτάρνετ και θα δώσουμε και το λόγο στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής μας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Σίτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι που δέχεστε την ε, πρόσκληση ε, την, που δέχεστε να παρέμβαση εδώ, η κυρία Μακταρνές, όπως είπε και ο Πρόεδρος, είναι συντονιστή για τη Μαυριτανία 2000. Πρόκειται για μια οργάνωση για τις γυναίκες που απασχολούνται στη μεταπληκτική βιομηχανία αλευτικών προϊόντων στη Μαυριτανία. Επίση, ε, είναι και μέλο ε, τη ΜΚΟ τη Μαυριτανία, Public What You Pay, και όπω ξέρετε, δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο θέμα τη διαφάνεια και προς αυτή την κατεύθυνση οι συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι σήμερα ήταν ε, ε ουσιαστικά θερμοί υποστηρικτές διαφανείς, αλλά θέλουμε να πάμε και πιο πέρα και θα δώσω αμέσω το λόγο στην κυρία Μκτανάκη για να κάνει μια παρουσίαση και κατόπιν οι συνάδελφοι μπορούν να τις θέσουν ερωτήσεις. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ιζαμπέλα, που μου έδωσε σε αυτή την ε, ευκαιρία να απευθυνθώ στην Επιτροπή Αλίας. Για μένα είναι πρώτη φορά που βρισκόμαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Μαυριτανία είναι μία από τις χώρες ε, που έχει ε, ουσιαστικά ε, πολύ μεγάλη δυνατότητα αλίας, αλλά όπου αλλιεύεται και πάρα πολύ ακτές της. Η πιο σημαντική, πιο σημαντικός τομέας μας είναι η αλία, όμως η αλία στη Μαυριτανία είναι για εξαγωγή. Υπάρχουν πάρα πολλές συμβάσεις στη Μαυριτανία, πολλές συμφωνίες, υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που αλλιεύουν στα πλαίσια συμφωνιών, όπως αυτές που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ελεύθερες συμφωνίες με Κίνα, Ρωσία, με διάφορες χώρες που έρχονται να αλλιεύσουν στη Μαυριτανία, δυνάμει κάποιες συμφωνίες. Αλλά υπάρχει μεγάλη διαφάνεια στις συμφωνίες αυτές, είτε είναι διμερείς, είτε είναι ελεύθερες συμφωνίες, ε, είτε ε, είναι στο πλαίσιο διμερούς ε, αδειοδότησης ή ελεύθερης αδειοδότησης. Όμως η δική μας επιθυμία ως οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που εργάζεται στον τομέα της αλίας είναι στο επίπεδο της, των συμφωνίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον να υπάρχει ένα πλαίσιο ναι, υπάρχει, μια διαδικασία της συμφωνίας αυτής ε, που γίνεται σε τοπικό επίπεδο, ενώ με συμφωνίες όπως έχουμε με την Κίνα, που είναι ελεύθερου τύπου, με ελεύθερες άδειε, ε, δεν ε, βλέπουμε τίποτα, τίποτα δεν ακούμε και πρόκειται για πλήρη αδιαφάνεια. Μία άλλη επιθυμία μας ως εκπρόσωπος της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα της αλίας είναι το εξή. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενθαρρύνει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη μια βιώσιμης ελεία στη Μαυριτανία και το πλαίσιο αυτό να είναι πολύ πιο γενικευμένο, να γενικευτεί ακόμη περισσότερο. Δηλαδή να μην αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ζητάμε γενικευμένη πρόσβαση σε επίπεδο διάφορων συμφωνιών και συμβάσεων με τη Μαυριτανία. Αρδράτω αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο για το ψήφισμα που ανέκρινε για τη Μαυριτανία, κυρίως ε, σε σχέση με τα άρθρα 12 και 14, σε σχέση με τη διαφάνεια, τη συμμετοχή της ε, κοινωνίας, ε, των πολιτών και των διάφορων πρωταγωνιστών και της προστασίας των πόρων. Αλλά θα θέλαμε το πλαίσιο αυτό να γίνει θεσμικό, δεν θα πρέπει η Μαυριτανία να μπορεί να πουλά τα ψάρια της στην Κίνα ε, με διαφορετικούς όρους και να χρησιμοποιείται διαφορετικό όρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρχει ένα γενικευμένο θεσμικό πλαίσιο για τη Μαυριτανία για να μπορέσουμε πράγματι να διαπραγματευτούμε ε, με ένα πολύ πιο κατάλληλο τρόπο για την εξαγωγή των ελευτικών μας προϊόντων. Η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση αξίζει αυτό που αξίζει, αλλά η συμφωνία με την Κινά είναι διαφορετική, γιατί στην περίπτωση εκείνη υπάρχει αδιαφάνεια. Ξέρουμε ότι η Βρυτανία πουλά τα ψάρια της στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο μιας συμφωνίας 4 ετών, ενώ για την Κίνα είναι 25 έτη. Για την Κίνα Η συμφωνία ισχύει 25 χρόνια. Και αυτό που προβλέπεται να κάνει είναι να γίνεται μια αναθεώρηση κάθε 5-6 χρόνια. Να, αλλά δεν υπάρχουν ε, φόροι, δεν ε, καθορίζονται οι συνθήκες εργασίας. Αυτό είναι καταστροφικό για τη Μαυριτανία. Έτσι λοιπόν ε, μια έκκληση γίνεται εδώ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο Επιτροπής Αλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Απευθύνω μια έκκληση ε, για να προσπαθήσετε να δείτε από κοινού με τη Μαυριτανία πώς μπορείτε να καταστήσετε αυτό το πλαίσιο θεσμικό έτσι ώστε οι συμφωνίες αυτές να εντάσσονται σε ένα κοινό πλαίσιο τουλάχιστον για να μην επιτρέπετε να κάποιοι να κάνουν ε, κάποια πράγματα τα οποία στους άλλους δεν επιτρέπονται. Γιατί όλα αυτά σημαίνουν απώλειες για τη Μαυριτανία. Και ξέρω ότι η Μαυριτανία από το 2005 προσχώρησε στην ε, πρωτοβουλία διαφάνειας για τις εξορροπτικές βιομηχανίες και από τότε δημιουργήθηκε μία επιτροπή στην ε, η οποία αποκαλείται «Δημοσίευστε αυτά που πληρώνετε» για να καταπολεμωθεί η διεθνή και από το 2005 προσπαθούμε να κάνουμε ένα μια έκκληση προκειμένου η Αλία να συμπεριληφθεί σε αυτές τις εξορρυκτικές βιομηχανίες, να θεωρείται ως εξορρυκτική βιομηχανία, για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε μηχανισμούς παρακολούθησης στη Μαυριτανία. Ε, δεν ε, υπήρξε συμφωνία για καταπολέμηση σε επίπεδο. Ε, μας είπαν ότι ε, αν τώρα μπούμε στο πλαίσιο της ελευθερικής Συμφωνίας θα πρέπει να υπάρχει μια παρακολούθηση θα πρέπει να διευρυνθεί η ε, των διαπραγματεύσεων και κατόπιν να δούμε και το δημοσιονομικό σκέλος. Ε, αυτό που θέλουμε εμείς να προωθήσουμε, αυτό που ζητάμε σε επίπεδο εθνικό είναι τουλάχιστον να συστηθούν κάποιοι μηχανισμοί διαφάνειας σε τοπικό επίπεδο και να τους υποστηρίξουμε εμείς με τη στήριξη των εταίρων μας ή με τη στήριξη των δωρητών. Αδράτω λοιπόν την ευκαιρία για να απευθύνω αυτή την έκκληση εδώ, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να εξετάσει και αυτή την πτυχή της διαφάνειας, να λάβει υπόψη αυτή την πτυχή της διαφάνειας που είναι σημαντική. Ίσως ε, θα μπορούσε να αποτελούσε μία αρχή. Δηλαδή οι χώρες, ε, οι εφοπλιστές ε, που έρχονται να ψαρέψουν στη Μαυριτανία τουλάχιστον να δηλώνουν τι έχουν πληρώσει. Γιατί αυτό είναι μια πολυτελεία για μας. Δεν ξέρουμε τι έχουν πληρώσει. Ε, και στο πλαίσιο τη Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσα έχει πληρώσει η κάθε χώρα δύναμη τη στάδη τη Δίνα Σύμβαση. Τι θέλουμε λοιπόν εμεί τώρα. Θέλουμε να υπάρχει αυτό το πλαίσιο διαφάνειας και στην αλία. Και θα θέλαμε κάτι τέτοιο να ισχύει όχι μόνο για τη Μαυριτανία, αλλά και σε διεθνές επίπεδο να προσπαθήσουμε να εμπλέξουμε το ΙΤΕ. Και... Euh, και να προσθέσω κάτι ακόμα. Υπάρχουν ε, διαπραγματεύσεις ε, για τις ποσοστώσεις, για τις απορρίψεις, για το στόλιο κτλ. Αλλά ξέρω ότι σε ό,τι αφορά τη Μαυριτανία στο πλαίσιο των συμφωνιών, των ελεύθερων αδειών, υπάρχουν πάρα πολλά παρεπιδόντα αλλιεύματα και πολλές απορρίψεις. Θέλουμε λοιπόν να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθήσει να γενικεύσει τις πολιτικές Λοιπόν, ξέρω ότι υπάρχουν και άλλε χώρε, ασιατικέ χώρε, χώρε από την Αμερική αλλά και ευρωπαϊκέ χώρε που αλλιεύουν στη Μαυριτανία. Πρόκειται λοιπόν για τι ίδιε χώρε ε, που ε, έχουν νομοθεσία στα δικά του εγχωρία. Θα πρέπει να σκεφτούν να το κάνουν και αλλού όμω αυτό. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι Ευρωπαίοι που θα έρθουν να αλλεύσουν στη Μαυριτανία. Ε, πέρα από ε, το πλαίσιο το οποίο έχει συσταθεί. Έχουμε και πλειοκτήτες, έχουμε και εφοπλιστές που προέρχονται από τις ίδιες χώρες, αλλά αλλιεύουν ακολουθώντας μια διαφορετική ηθική. Έτσι λοιπόν θέλω να επιστήσω εδώ την προσοχή σας σε αυτό το θέμα, για να το σκεφτείτε. Ίσως ε, μπορείτε να πείτε ότι δεν μπορούμε να μπλακούμε στην πολιτική των άλλων, μιλάμε για εθνική κυριαρχία των χωρών. Αλλά ξέρετε, πολλέ φορές οι αναπτυσσόμενε χώρες ακούν πολύ περισσότερο τους δωρητέ τους παρά τους δικούς τους ε, υπηκόους, παρά τις δικές τους οργανώσεις, του δικού τους ε, πρωταγωνιστές στον κλάδο. Εμείς θέλουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας βοηθήσει μας ως ε, πρωταγωνιστές επιτόπου για να πάρουμε μέτρα. Γιατί όταν αυτά τα μέτρα ε, ζητούνται από το εξωτερικό, η ανταπόκριση είναι μεγαλύτερη. Θέλουμε λοιπόν να πάμε στο δυνατόν μακρύτερα. στα πλαίσια αυτή τη μάχη, για να προσπαθήσουμε να έχουμε το των δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα και προκειμένου η Αλία στη Μαυριτανία να είναι πολύ πιο βιώσιμη, για να διατηρούνται οι πόροι και να είναι και πιο αποδοτική και για τους πολίτες αλλά και για τους εισαγωγείς. Γιατί αν δούμε τι συμβαίνει σε επίπεδο το 99% της παραγωγής είναι για εξαγωγή. Δεν υπάρχουν βασικές υποδομές, ε, δεν υπάρχουν επενδύσεις, δεν υπάρχει αποδοτικότητα του τομέα και δεν υπάρχει ε, θετική, θετικό όφελος για τους πολίτες από τις επενδύσεις αυτές από τις ελευτικές δραστηριότητες. Θέλουμε εμείς λοιπόν διαφάνεια γιατί και στο επίπεδο της διατήρησης των πόρων πρέπει να προσδώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Μοντάρ που ήρθατε από τόσο μακριά για να μας κάνετε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα και ενημερωτική παρουσίαση. Θέλει η κυρία Λέβιν ε, να προσθέσει κάτι πριν ακούσουμε την Επιτροπή. Η κυρία Φράγκα. Eh, Ευχαριστώ την προσκεκλημένη μας ε, για όσα μας είπε γιατί ξέρετε ότι τίποτα δεν μας εκπλήσει στο πλαίσιο της Μαυριτανίας όταν οι κυβερνήσεις δεν είναι διαφανείς, δεν είναι διαφανείς με κανένα και το πρόβλημα δεν είναι ότι εμείς μπορούμε να το λύσουμε γιατί αυτοί έχουν την εθνική κυριαρχία ε, για να πούν τι κάνουν ή τι δεν κάνουν. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθεί να μάθει ποιοι άλλοι αλλιεύουν, πώ αλλιεύουν και τι για να υπολογίσουμε τα πλεονάσματα. Ναι, αυτό γίνεται, αλλά κατά τα λοιπά αυτή είναι αρμοδιότητα της κυβέρνηση τη Μαυριτανίας. Εμείς μπορούμε να υποστηρίξουμε και να πούμε ότι θέλουμε μεγαλύτερη διαφάνεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρκετή διαφάνεια, τουλάχιστον οι ε, συμφωνίες όλες δημοσιεύονται επισήμως. Όμως αυτό που ε, την προσοχή μα, είναι, που προκαλεί την προσοχή μα, είναι ότι η κυβέρνηση Μαυριτανίας με άλλες χώρες όπως Ρωσία, Κίνα κτλ. έχει συνάψει συμφωνίες 25 ετών υπό υπόπτε συνθήκες πολλές φορές. Ενώ με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τώρα εμπλοκή της συμφωνίας. Ε, οι απαιτήσει ε, κυρίως για τις τρεις κατηγορίες ελίας που χρησιμοποιούν πλήρως συμφωνία είναι αδύνατο να πληρωθούν. Υπάρχουν ε, τομεί, υπάρχουν κλάδοι που μπορεί ότι δεν θέλουν συμφωνία με τη Μαυριτανία και εγώ θα ήθελα να ξέρω βάσει αυτού τι σκέφτεται η προσκεκλημένη μας. Εγώ σας είπα ότι έχω συμμετέχει σε ε, συναντήσεις ε, με εκπροσώπους του κλάδου και κάποιοι είπαν ότι δεν θέλουν συμφωνία με τη Μαυριτανία γιατί οι απαιτήσει είναι τέτοιες που τελικά δεν μπορούσε να ενδιαφέρουν η συμφωνία. Έτσι λοιπόν, ε, τώρα έχουμε κάποιες κυβερνήσεις τρεις χωρών που δίνουν προτεραιότητα σε στόλους, ε, που αλλιεύουν ε, με λιγότερους περιορισμούς από ό,τι ο στόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελικά ευνοούνται οι στόλοι αυτοί. Γιατί? Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε και για διαφθορά και για άλλα θέματα που δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε. Αλλά σίγουρα κρύβονται από πίσω. Τώρα αυτά που είπε πιο συγκεκριμένοι μας για τις απορρίψεις ε, και τα λοιπά, ότι δεν ε, μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε μόνο πόρους, αλλά θα έπρεπε να υποστηρίξουμε και την ανάπτυξη επιτόπου. Εγώ πιστεύω ότι ο ευρωπαϊκός ε, τομέας έχει συμφέρον και στη συγκεκριμένη περίπτωση της Μαυριτανίας, γιατί έχουμε τον πελογικό στόλο, ο οποίος πραγματικά έχει κάθε συμφέρον να μπορέσει να επενδύσει εκεί. Και το ξέρω γιατί έχω μιλήσει με τους πλειοκτήτες, με τους εφοπλιστές. Το πρόβλημα που έχει η Μαυριτανία είναι ότι τα κονδύλια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που δίνουν άλλες χώρες για την ανάπτυξη του ελευτικού τομέα στη Μαυριτανία και των υποδομών ίσως δεν χρησιμοποιούνται έτσι όπως θα έπρεπε. Λογικά για να για να έχουμε ανάπτυξη επιτόπου πρέπει να υπάρχουν κάποιες ελάχιστες υποδομές και αυτό πρέπει να γίνει με την βοήθεια της ε, κυβέρνηση Μαυριτανία Τώρα και το λιμάνι του που είναι το πιο σημαντικό κειμένο, ακόμη και εκεί έχουν προβλήματα να μπουν τα σκάφη και δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα αυτά, δεν ε, ε, έχουν λυθεί τα προβλήματα του λιμένα. Αυτό φυσικά είναι πρώτερη προϋπόθεση προκειμένου ο κλάδος να μπορέσει πράγματι να αναπτυχθεί σημαντικά στα λιμάνια. Ε, και πραγματικά ε, Σα είπα ότι επειδή μιλώ εγώ με εκπροσώπου του κλάδου, επιθυμούν κάτι τέτοιο. Τώρα, η κυβέρνηση Μαυριτανία έχει δυσκολία για να δαπανίσει την ε, συμφωνία τις ενισχύσεις που λαμβάνει, ίσως θα μπορούσε να δώσει προσθεμένη αξία στην ανάπτυξη του αλληλευτικού κλάδου στη Μαυριτανία. Πάντως, εγώ θα ήθελα ε, να μας πείτε τι σκέφτεστε στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν καν να υπάρχει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κυρία Γκαρσία Γέρο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστούμε για τις ε, πληροφορίες που μας δώσετε για το τι συμβαίνει στη χώρα σας και για το τι συμβαίνει σε μια κατάσταση νομίζω ότι ε, κάποιοι άλλοι καθορίζουν τις συνθήκες ε, και η Μαυριτανία τις δέχεται. Και όπως είπατε και εσείς υπάρχει τεράστια διαφάνεια. Και βέβαια ίσως να υπάρχουν ε, και άλλες ε, καταστάσεις που εγώ δεν θα αναφέρω τώρα εδώ, γιατί θέλω να είμαι σόφρον. Όμως ε, αυτά που εμείς ε, θέτουμε στην ε, πολιτική μας για τη βιώσιμη αλία και τη μεταρρύθμιση που πηγαίνει και πιο πέρα και μιλάμε και για τον κώδικα δεοντολογίας, ε, όχι μόνο για κώδικα νομικό, περιβαλλοντικό, αλλά λαμβάνουμε υπόψη και ε, αν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατικές ελευθερίες, για όλα αυτά πρέπει να κάνουμε μία προσπάθεια. Εμείς ίσως από εδώ δεν μπορούμε να πάμε πιο πέρα από το να απαιτήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Συμβούλιο, από την Κομισιόν να δημιουργήσει ένα μόνιμο διάλογο προκειμένου να είναι δυνατόν ε, να, έχουμε αυτές τις διμερείς συμφωνίες ε, και να μας οδηγούν στο εξή. Αν έχουμε ένα εταίρο τόσο μεγάλο εταίρο όπως η Κίνα, να μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα, γιατί δεν πρέπει μόνο να μιλήσουμε με τη Μαυριτανία για να δούμε τι συμβαίνει και γιατί παρουσιάζονται τόσε δυσκολίε ε, για τη σύναψη συμφωνία. Φυσικά, αν ε, η Κίνα προσφέρει τόσα μεγάλα πλεονεκτήματα και αν δεν υπάρχει κανένα ε, έλεγχο, αν δεν τίθεται καμία προπόθεση για τι δημοκρατικέ ελευθερίε, για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για το σεβασμό του περιβάλλοντο κτλ., τότε πράγματι μιλάμε για δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή δεν μπορούμε ε, μια φιλοσοφία ή ένα πολιτικό σχέδιο να το προωθούμε μεν και από την άλλη ε, στην αγορά να κινούμαστε χωρίς να υπάρχει κανένας περιορισμός και αυτό συμβαίνει και το επιτρέπουμε και στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιτρέπουμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή εμείς ε, συστήνουμε στη Μαυριτανία και τη λέμε πρέπει να κάνετε αυτά, αλλά δεν κάνουμε τίποτα για την Κίνα. Για να απαιτήσουμε από τη Μαυριτανία να πληρεί κάποιε προποθέσει, πρέπει να απαιτήσουμε και από την Κίνα και από όλε τι χώρε που δεν πληρούν τι προποθέσει αυτέ, που δεν σέβονται, ε, να σεβαστούν του ίδιου κανόνε του παιχνιδιού, γιατί αυτό πηγαίνει πιο μακριά από το θέμα τη εθνική κυριαρχία. Νομίζω ότι είναι ηθικό το ζήτημα, είναι θέμα υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ναι, μπορούμε να μιλήσουμε για την αλία, αλλά νομίζω ότι εδώ είναι σημαντικό αυτό το θέμα, γιατί όπως είπατε και εσείς, ε, ε, έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της ε, παραγωγής, το οποίο στη συνέχεια εξάγεται και εμείς δεν ξέρουμε ποιες προϋποθέσεις. Έτσι λοιπόν εμείς επειδή ε, έχουμε πολύ μεγάλες εισαγωγές θέλουμε να ξέρουμε τι καταναλώνουμε γιατί μας ενδιαφέρει και η υγεία των πολιτών. Εσείς ε, έχετε, όχι, έχετε την ηθική, όχι μόνο την πολιτική δύναμη, να έρχεστε εδώ να μας ζητάτε μέσα στο όριο που έχουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εγώ δεν ε, ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει, σε ποιο άλλο πλαίσιο, πέρα από αυτά που είπα σήμερα, αλλά ξέρω τι πρέπει να κάνουμε και ότι πρέπει να σας ε, υποστηρίξουμε και εσάς και τις υπόλοιπες χώρες Και εφόσον ε, υποστηρίξαμε κάποια στιγμή να, να μπορούν να βγαίνουν οι άνθρωποι στον δρόμο για να ζητήσουν ελευθερία και δημοκρατία, τι άλλο να σας πω εδώ, μπορώ να σας πω, δεν θα σας πω τίποτα άλλο, παρά το ότι εδώ και ως γυναίκα βλέπω ότι σε αυτές τις χώρες, παρόλο που γίνεται προσπάθεια να κλείσουν τα στόματα, και παρόλο που προσπαθούν ε, να σας κάνουν να μην μιλάτε τελικά εσείς οι γυναίκες ε, υψώνετε τη φωνή σας και έχετε ηγετική θέση και θέτετε τα διάφορα προβλήματα επιτάπητος. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν και πραγματικά η Ισπανική Αντιπροσωπεία, του σοσιαλιστές σε ό,τι μπορεί θα σας βοηθήσει. Είμαι στη διάθεσή σας. Ευρωπαϊκής ε, Θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου που σας γνώρισα και θέσατε με εξαιρετικό τρόπο διάφορα σημαντικά ζητήματα. Ε, κοιτάξτε, υπάρχει ένα ψήφισμα που εγκρίθηκε στο Κοινοβούλιο, ε, που πραγματευόταν σχετικά ζητήματα και μας λειτουργεί ως ε, ε, κατευθυντήρια γραμμή για την περαιτέρω δράση μας στη Μαυριτανία. Δείτε τι περιέχει αυτό το ψήφισμα και έχω αποσπασματικά, έχω φτιάξει ένα πάτσουρ από διάφορα αποσπάσματα του ψηφίσματος για να τα συσχετήσω με τις δικές σας παρατηρήσεις. Θα δείτε λοιπόν ότι στο μέτρο που μιλάμε για κατευθυντήριε ε, γραμμέ, αυτό που ζητήσατε εσείς είναι κάτι ε, στο οποίο αποσκοπούμε ούτω ή άλλω. Κατά τα λοιπά, ε, οι αρχές που προτείνεται να εφαρμόσουν μας βρίσκουν σύμφωνους ε, ως προς την μελλοντική μεταρρύθμιση εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και στις εξωτερικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης επικρατούν αυτές οι αρχές όπως βλέπετε και στην ανακοίνωση περί των αρχών που διέπουν οποιαδήποτε μεταρρύθμιση των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης και στη συγκεκριμένη περίπτωση της Μαυρετανία, δίκιο έχετε, συνεχίζονται διαπραγματεύσεις. Φυσικά δεν αρκεί να ζητήσουμε τη συγκατάθεση του, ε, της κυβέρνησης της Μαυρετανίας θα δούμε τι θα γίνει με τις διαπραγματεύσεις. Η διαφάνεια πάντως για θέματα όπως η στόλη είναι κάτι που ζητούμε ρητά από την κυβέρνηση, αλλά είναι λίγο δύσκολο να σας πω περισσότερα πράγματα τώρα. Ε, για τα ποσά Συνεχίζουμε τις προσπάθειες. Ε, πάντως, ε, για λόγους διαφάνειας θα υπάρξουν επίσημοι λογαριασμοί, ε, θα υπάρχει σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό και άρα μπορεί το Κοινοβούλιο να παρακολουθήσει τους εθνικούς λογαριασμούς και να δει ποια ακριβώς είναι τα ποσά που εισπράττει η κυβέρνηση. Φυσικά θα μεριμνήσουμε ώστε να επικρατήσει διαφάνεια και για τις τεχνικές προδιαγραφές και θα είναι διαθέσιμη τεκμηρίωση από τη στιγμή που θα καταλήξουμε σε συμφωνία και μετά. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν αυτές τις ε, αρχές ε, που προτείνουμε, ε, πρώτη μας βασική μέρη να είναι να μπορεί να αλλιεύει και ο εγχώριος στόλος, αλλά φυσικά και ο στόλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν γίνει δεκτή η συμφωνία, η Μαυριτανία θα έχει στη διάθεσή της εργαλεία για να εκπονήσει ε, ε, πολιτική, θα έχει και ε, τα απαιτούμενα οικονομικά μέσα για να καταρτήσει μια εθνική πολιτική. Είμαστε πολύ πιο διαφανείς από όλους τους υπόλοιπους παίκτες εισαγωγικά σε αυτή την αρένα. Και αυτό βάσει των ε, κατευθυντηρίων που βλέπετε στο ψήφισμα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις. Σα ευχαριστούμε κύριε Πτυμπέρ. Κυρία Μόκτα, θέλετε μήπω να απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα της ε, συναδέλφου κυρία Φράγκα. Σε σχέση με τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα σας πω ακριβώς ποια είναι η θέση μας. Επειδή δραστηριοποιούμαστε στον αλλιευτικό κλάδο όλος ιδιαίτερος και στα πλαίσια της συμφωνίας ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα σας έλεγα ότι υπάρχουν ε, και ρυθμιστικές διατάξεις και συμφωνία ήδη ε, η κοινωνία των εταίρων ε, είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Το κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα του κλάδου, τη διατήρηση των αποθεμάτων κτλ. Ε, στην Κίνα δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, παραδείγματος χάρη. Είναι εντελώ διαφορετική κατάσταση στη Μαυριτανία. Αυτό που θέλουμε εμεί είναι, επιθυμούμε μάλλον διακαώ την υπογραφή Τη συμφωνίας. Έχει περιορισμού συμφωνία, αλλά έχει και πλεονεκτήματα. Ιδού η τρανή απόδειξη υποφαινόμενη. Έρχομαι εδώ στο Κοινοβούλιο να εκφράσω την άποψή μου. Στην Κίνα δεν με καλέσανε ε, και σε αυτές τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου δεν ξέρουμε τι κρύβεται πίσω, δεν γνωρίζουμε τα ποσά, δεν γνωρίζουμε την ε, χρηματοδότηση, δεν ε, έχουμε λέγην. οπότε σε σχέση με την συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό το ζητάμε συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Θα θέλαμε να μάθουμε, ε, να συνειδητοποιήσουμε μάλλον ότι ψαρεύουμε τον ίδιο ωκεανό, τα ίδια ψάρια ψαρεύουμε, άρα δεν μπορούμε να τα πουλάμε σε διαφορετική τιμή και να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ε, βεβαίως ε, θα είναι πιο ζημιογόνος αν θέλετε η, συμφωνία για μας από ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ε, πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειε η δική μας η κυβέρνηση ούτω ώστε να... είναι θεσμικά στεγανό το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων στο μέλλον. Επίσης να εμπλακούν ε, όλοι οι εταίροι στις διαπραγματεύσεις γιατί οι πιοφουσιολογικές συνθήκες γίνονται διαπραγματεύσεις και κλεισμένων των θυρών. Ξέρετε, ορισμένες φορές εμπλεκόμαστε αλλά με την ιδιότητα του παρατηρήτη. Άρα δεν λαμβάνεται η ε, υπόψη η θέση μας. Δεν ακούγεται η άποψή μας αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ε, προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήθελα να πω τα εξή ε, για τους οικονομικούς πόρους. Θα σας εξηγήσω ότι στην Μαυριτανία ε, έχουν διοχετευτεί κάποια κονδύλια αλλά δεν επανεπενδύθηκαν ποσά στον τομέα της αλίας. Δηλαδή, εμείς ζητάμε ρήτρα παρακολούθησης των συμβάσεων. Εγώ, παραδείγματο χάρη, συμμετέχω στην αξιολόγηση των συμφωνιών. Η Μαυριτανία δεν τήρησε τις ρήτρες της συμφωνίας εδώ και χρόνια προσπαθούμε ε, να αλλάξουμε την κατάσταση. Παρόλα αυτά υπογράφονται συμφωνίες με τη Μαυριτανία. Δηλαδή πρέπει να προβλέπετε ρήτρα τήρησης ε, των ε, συμβάσεων, γιατί αλλιώς θα είναι μεγάλες οι ζημιές. Ξέρω ότι υπάρχει χρηματοδότηση για τι υποδομέ από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμία υποδομή δεν έχει δημιουργηθεί νέα. Παρόλα αυτά έχουν υπογραφεί οι συμφωνίε. Ζητώ λοιπόν να ε, καταστήσουμε γενικότερο το πλαίσιο, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε έναν ε, ε, εποπτικό μηχανισμό, έναν μηχανισμό παρακολούθηση για να υποχρεωθούν οι τρίτες χώρες. Φυσικά είναι θέμα κυριαρχίας, εθνικής κυριαρχίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά την φύση της κυβέρνησης της Μαυριτανίας. Αλλά ξέρετε ότι θα μας σας ακούσουν εσάς περισσότερο από ότι εμάς. Εσείς πληρώνετε, εσείς δίνετε κονδύλια, οπότε θα σας ακούσουν πολύ περισσότερο. Θα ακούσουν περισσότερο δηλαδή σε εκπροσώπους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ότι τον ντόπιο πληθυσμό. Μόνο αυτό σας ζητάμε. Σας ευχαριστούμε κυρία Μοντελέο, κύριο Στίβενσον. Δεν έχουμε χρόνο, Ιζαμπέλα. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις ε, κάτι τελευταίο. Όχι. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και πάλι από πλευρά τη Επιτροπή την κυρία Μόρτα που γιατί ήταν πραγματικά εξαιρετική, πολύ ενδιαφέρουσα ε, η παρουσίαση του ζητήματο ε, και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη ε, πολλά από τα στοιχεία που μα δώσατε. Λοιπόν, στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μα θα δώσω το λόγο στον ε, κύριο Φερέιρα για το σχέδιο έκθεσης ε, για τη μεταρρύθμιση κοινή αλληλευτικής πολιτικής ε, και την αλληλεία μικρής κλίμακος. Καρκινοβατούμε τώρα, γυρίσαμε στο 14. Συγγνώμη πρόεδρε για την καθυστέρηση, αλλά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος έπρεπε να συζητήσουμε κάποια θέματα για την αλληλεία και ακριβώ υπήρχε και μια γνωμοδότηση για την ΚΟΑ. Θέλω να ευχαριστήσω την Ιζαμπέλα για την δυνατότητα ανταλλαγή των ε, σημείων. Εμεί. κάναμε ήδη ε, μια πρώτη συζήτηση για το θέμα αυτό. Βέβαια δεν είχαμε το γραφείο εργασία. Είναι οργανωμένο σε τέσσερα κεφάλαια. Το προ, στο πρώτο γίνονται ορισμένε γενικέ ε, ε σκέψει για τον ορισμό τη αλληλεία μικρή κλίμακα, δηλαδή τι είναι η μικρή παράκτεια αλία και αλία στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία ανάλυση του αντικτύπου των διάφορων νομοθετικών εργαλείων που συζητούμε είτε του γενικού κανονισμού είτε του κανονισμού για την ΚΟΑ είτε της πρότασης κανονισμού για το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας, ποιος είναι ο αντίκτυπος αυτών των τριών νομοθετικών μέσων ε, στην αλία μικρής κλίμακας. Και το τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται κάποιοι γενικοί προσανατολισμοί και κάποιες προτάσεις συγκεκριμένες για το πώς ε, θα πρέπει να αξιολογηθεί και να δοθεί νέα αξία στην αλία μικρής κλίμακας και ε, πώς ε, θα αναγνωρίσουμε την αξία της, κάτι που δεν γίνεται δυστυχώς στις προτάσεις της Κομισιόν. Οι, οι προτάσεις της Κομισιόν ιδιαίτερα ανεπαρκή τρόπο χειρίζονταν ε, την ε, ε, αλία μικρής κλίμακας σε αυτά τα δύο τελευταία κεφάλαια, στο τρίτο και στο τέταρτο, έχουμε προτάσεις, συστάσεις που ο καθένας από τους δύο εισηγητές μπορούν να λάβουν υπόψη στο έργο τους. Δεν θα αναφερθώ εδώ εξαντλητικά, απλώς θα αναφερθώ σε μια-δυο, αλλά πολύ σύντομα γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Εγώ θα ήθελα να σας ακούσω βασικά. Προτείνεται ένας νέος ορισμός για την αλία μικρής κλίμακας ε, που διορθώνει τον περιοριστικό ορισμό που υιοθετεί η Κομισιόν στις ε, προτάσεις της. Η Κομισιόν λέει ότι είναι δύσκολο να λάβουμε υπόψη άλλα κριτήρια. Είναι ε, δύσκολο να έχουμε υπόψη μερικά κριτήρια παρά μόνο ένα, όμως ε, κοιτάξτε, οι ε, που προ... οι... οι που προκύπτουν από το να έχουμε ένα περιοριστικό ορισμό είναι πολύ μεγαλύτερες από το να έχουμε ένα πιο διευρυμένο ορισμό. Έτσι λοιπόν προτείνω εγώ εδώ κάποιε τροποποιήσει σχετικά με τον ορισμό στην πρόταση και έχουμε και το θέμα της διαχείρισης της εγκύτητας και στο ότι ε, στην μεταρρύθμιση πρέπει να προωθήσουμε περισσότερο την περιφερειοποίηση και το θέμα της εγκύτητας. Πρέπει να πάμε πιο μακριά από αυτό μας προτείνει η Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη Γνωρίζουμε ότι διαφέρει η πραγματικότητα τη αλίας αλλά και τη Αλία μικρή κλίμακα στα διάφορα κράτη-μέλη από το βορρά στο νότο και πρέπει να δώσουμε επαρκή ευελιξία στα κράτη-μέλη προκειμένου να μπορέσουν να υπερασπίσουν και να δώσουν αξία στο ρόλο αυτό το με τώρα για τις μεταβάσιμε ελευτικές παραχωρήσεις θα πρέπει να μην υπάρχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, δεν θα πρέπει να επιβάλλεται υποχρεωτικά ένα σύστημα σε όλα τα κράτη-μέλη δεν ε, θα αναπτύξω εδώ τα επιχειρήματά μου γιατί το έχω κάνει σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν. Όμως εμείς πέρα από την ποσότητα του στόλου πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ποιότητα του στόλου. Έχουμε διάφορες εμπειρίες και εδώ απευθύνουμε κυρίως την κυρία Ρόντουστ που είναι η συγγήτρια για το βασικό κανονισμό. Έχουμε διάφορες εμπειρίες εφαρμογής ε, των παραχωρήσεων, μεταβάσεων παραχωρήσεων που οδήγησαν στον αριθμό, σε, σε, μείωση του αριθμού των σκαφών, αλλά φυσικά αυτό δεν σήμανε πάντα ότι είχαμε και μείωση της ελευτικής προσπάθειας. Έτσι λοιπόν αυτοί που έμειναν τελικά αλλιέυαν περισσότερο και αυτοί που έφυγαν τελικά πήγαιναν αλλού να αλλιεύσουν. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι η προσέγγιση που υιοθετείται εδώ ε, δεν είναι σωστή και δεν μπορούμε να το εγγλήσουμε. Εμείς πρέπει να λάβουμε υπόψη στην ποιότητα και όχι μόνο την ποσότητα. Και ε, όπως προτείνει η Κομισιόν, αν εφαρμοστεί το σύστημα των μεταβάσιμων συλλεκτικών παραχωρήσεων έτσι, έχουμε μείωση του στόλου, αλλά δεν ε, αποσύρονται ε, τα σκάφη που είναι τα πιο ζημιογόνα. Το αντίθετο μάλιστα από την οικονομική σκοπιά θα σταματήσουν να δραστηριοποιούνται τα σκάφη τα πιο ευπαθή. Και αυτό είναι ένα άλλο σημείο που αναφέρεται εδώ, δηλαδή Έχουμε και κάποιες προτάσεις ε, από τον κύριο Στίβενσον να λάβουμε υπόψη αυτές τις ε, ιδιαιτερότητες της ε, μικρής αλίας σε περιβαλλοντικό και σε κοινωνικό επίπεδο και θα πρέπει το Ταμείο να δημιουργήσει το δικό του ρόλο, θα πρέπει να δημιουργήσουμε τα μέτρα που να μας επιτρέπουν να γνωρίσουμε αυτούς τους εξωτερικούς παράγοντες, τους θετικούς προτείνεται ένα κοινοτικό πρόγραμμα στήριξης ε, στην ε, αλία μικρή κλίμακα και από τον κύριο Καντέκα έχουν γίνει κάποιε προτάσει για να ληφθούν ε, υπόψη, ε, μάλλον έχουν γίνει στον κύριο Καντέκα κάποιε προτάσει για να ληφθούν υπόψη στην γνωμοδότηση για το ΕΤΘΑ. Η στήριξη στη μικρή Ελία δεν αντίκειται της ε, πρόταση Μπορούμε να εγγυηθούμε κάποιου ελέξεις τους πόρους για αυτά τα τμήματα του στόλου, το θέμα της ανανέωση του τομέα ε, προτείνεται ανανέωση του τομέα τη διδοκαλλιέργεια. Δεν είναι δυνατόν να το κάνουμε αυτό χωρί να το προτείνουμε και για την αλία μικρή κλίμακα. Πρέπει να προσδώσουμε αξία και στο ρόλο των γυναικών στη μικρή αλία. Επίσης γίνονται κάποιες σκέψεις σχέση με την χρήση τη αποκλειστική οικονομική ζώνης ε, ε, και έχουμε θετικές επιπτώσεις που πρέπει να αναπτυχθούν, πρέπει να δοθεί δυνατότητα στα κράτη-μέλη να πάνε παραπέρα από τα σημερινά 12 μίλια, κυρίως ε, στις άκρως απομακρυσμένε περιοχές. Πρέπει να εξεταστεί δυνατότητα να φτάσουμε μέχρι τα 200 μίλια και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μπορούν να λάβουν μέτρα προστασίας, διατήρησης, ε, μέτρα ε, κατά του κατακαιρματισμού για να έχουμε κάποιες περιοχές όπου θα μπορούν να αλλιεύουν οι μικροί αλλοί. Και εδώ έχετε ένα παράδειγμα αυτής του κατακαιρματισμού στο χώρο που εγγυάται προτιμητέα πρόσβαση ε, στο στόλο που είναι πιο συνδεδεμένος με τις ε, παράκτης κοινότητες. Επίσης προτείνονται κάποιοι μηχανισμοί έκτακτου ανάγκης ε, καθώς αυτά τα τμήματα του στόλου υφίστανται πιο αρνητικές συνέπειες από εξωτερικά σοκ από ό,τι πιο ανταγωνιστικά τμήματα του στόλου προτείνονται κάποιοι μηχανισμοί που να μπορούν να λειτουργούν σε έκτακτες ε, περιπτώσεις, σε έκτακτες Δεν υπάρχει κατέφυγη και πρέπει να το σκεφτούμε στη μελλοντική μεταρρύθμιση. Από μένα αυτά και θα ήθελα τώρα να ακούσω τις δικές σας συνεισφορές. Can I say I've got... Ευχαριστούμε πολύ. Εφτά συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο και έχουμε 9-10 λεπτά μέχρι το, τη λήξη της συνεδρίασης. Με το ρολόι λοιπόν, ένα λεπτό ο καθένας, γιατί έχουμε και την Κομισιόν και τον ε, ε, κύριο Φερέιρα ε, να ακούσουμε. Στην επόμενη συνεδρίαση μπορούμε να επανέλθουμε. Τώρα όμως δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τις 12.30 πριν διακόψουμε. Κυρία Φράγκα. Κοιτάξτε, σε ένα λεπτό δεν μπορώ να πω τίποτα. Απλώ Ήθελα να πω για την γνωμοδότηση του κύριου Φεραίρα ότι έχει μια εντελώ ειδηλιακή εικόνα για την μικρή παρακταλία. Δεν ε, είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα. Ε, εγώ θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για μια αλεία που δεν είναι τόσο κεφαλοποιημένη και έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο ε, στην επικράτεια και γι' αυτό πάντοτε μιλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θετική ενίσχυση όμως, ε, κοιτάξτε, ε, υπάρχουν και κάποια αρνητικά, δηλαδή πρέπει να έχουμε και υπόψη και τον αντίκτυπο που έχει στο οικοσύστημα, γιατί οι μικροί ελίες πάντοτε αλλιεύουν ε, στα πιο ευπαθή οικοσυστήματα που είναι κοντά στην εκτήση και για τις ITQs, για τις μονομένες ποσοστώσεις, ατομικές ποσοστήσεις. Δεν ξέρω γιατί επιμένετε τόσο πολύ. Όταν στην Πορτογαλία έχουμε πάνω από το 80% όπου δεν θα εφαρμοστεί, ενώ στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω το 70% ε, στο οποίο δεν θα εφαρμοστούν αυτέ τι ποσοστώσει. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλέ πτυχέ που θα θέλαμε να συζητήσουμε, αλλά εδώ δεν μπορούμε να συζητήσουμε τίποτα. Και τι κάνουμε, τελικά δεν μπορούμε να πούμε αυτά που σκεφτόμαστε. Thanks very much for that. Mr. Uh, one minute, please. Κοιτάξτε, δεν με έχω... Ε, πυρίλιο, πυρίλιο λέγομαι. Λέτε το όνομά μου στα ισπανικά. λοιπόν, σας ευχαριστώ. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Φερέιρα σχεδόν 100% και τον συγχαίρω για το έργο του. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κάποια προσπάθεια όμως περαιτέρω. Κοιτάξτε, εγώ προέρχομαι από μια τελική περιοχή που είναι παράκτια και έχω γνώση αυτών των θεμάτων. Ε, και μικρή αλία Δυστυχώ είναι σε δύσκολη κατάσταση, δεν υπάρχει δυνατότητα να βελτιώσουμε τις συνθήκες και Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να εξεύρουμε και άλλου μηχανισμούς που να είναι ικανοί να δώσουν μια όθηση σε αυτή την αλία μικρής κλίμακας, Μπαράκτη αλία. Κάτι τελευταίο. Ίσως δεν χρειάζεται να το πω, όμως σε ό,τι αφορά τα εχθίδια. Υπάρχουν ε, διάφορες ε, θέσεις, υπάρχουν και βιολόγοι οι οποίοι ε, κάνουν μια σειρά αξιολογήσεων για τα εχθίδια και θα ήθελα στο μέλλον να συζητηθούν αυτά. Ευχαριστώ. Oh, uh, next we have Mrs. κυρία τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Φερέιρα για την έκθεση. Συμφωνώ απόλυτα ότι η ποιότητα των στόλων είναι πολύ σημαντική και ότι πρέπει να δώσουμε προτιμησιακή πρόσβαση ε, σε αυτούς που είναι εντάξει βέβαια. Ε, δίκιο έχει και η κυρία Φράγκα που λέει ότι δεν είναι ότι η μικρή αλληλεία δεν βλάπτει ποτέ το περιβάλλον και δουλεύει και σε ευα... λειτουργεί, δραστηριοποιούνται και σε ευάλωτες περιοχές. Στις Αζόρες έχουμε υφαλοκρηπίδα πολύ περιορισμένη και είναι η αλληλιά σε ανοιχτή θάλασσα. Σε βάθος 40 μέτρων όμως ο αντίχτυπος είναι πολύ μεγάλος. Επίσης ε, για τα σκάφη μικρότερα από 10 μέτρα που δεν χρειάζεται να έχουν ημερολόγιο σκάφους ε, με βάση τον παρόντα κανονισμό. Ε, και αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε. Ευχαριστώ, κύριος Μπέσσερ. Σε ένα λεπτό, όπως είπε και η κυρία Φράγκα, τι να προλάβω να πω, είναι αδύνατον ε, να καλύψω όλες επιμέρους πτυχές αυτού του τόσο σημαντικού ζητήματος, επικροτώ τον κύριο Φερέιρα, διότι ρίχνει το φως της δημοσιότητας σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Η έκθεση είναι καλά ισοσκελισμένη, αλλά υπάρχει ένα θέμα μεθόδου εκπόνησης και προσανατολισμού της πολιτικής. Ε, ε τώρα, επειδή δεν έχω χρόνο, θα τα σχηματοποιήσω όλα. Ε, προτείνεται, κύριε Φερέιρα, να ε, διαφοροποιήσουμε στο μέγιστο ε, την μεταχείριση, δηλαδή να λαμβάνουμε υπόψη το οικονομικό, κοινωνικό προφίλ των περιοχών για να πάρουμε τις αποφάσεις και να θεσπίσουμε ειδικά καθεστώτα στον τομέα της αλίας, πολλαπλασιάζοντας τα διαφοροποιημένα μέτρα και η Ρίστο εμπαρόδο συμφωνούμε με τα μέτρα, ε, αλλά ε, προτείνεται κλαδικές εξαιρέσεις. Ε, εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται μία άλλη μέθοδος ώστε να ανακάμψει ο κλάδος. Δηλαδή, ε, πέρα από τα συντεχνιακά συμφέροντα, ποιο είναι το κοινό καλό ε, είτε μιλάμε για την μικρή αλία, για την παράκτη αλία, την εραστεχνική αλία, το βασικό κριτήριο κοινό ε, παρονομαστή είναι η επίτευξη τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση ε, που συνιστά προτεραιότητα για το μέλλον. Ακόμη και για την ε, μικρή παράκτη αλία, ζητώ συγγνώμη, δεν, δεν προλαβαίνω να αναπτύξω περαιτέρω τη θέση μου. Σα ευχαριστούμε κύριε Μπέσε. Τώρα δε πώ θα χωρέσετε όλοι, δυσκολευόμαστε. Τέλο πάντων, πέντε λεπτά έχουμε κυρία Ρόντου. Ευχαριστώ. Θα τα πω γρήγορα. Καταρχήν ε, συγχαρητήρια για την ενδιαφέρουσα έκθεση. Κάποια στιγμή ε, στο μέλλον ελπίζω να τα πούμε περισσότερο λεπτομεριακά. Ο ορισμός της μικρής αλίας στο βασικό κανονισμό το αμφισβητώ και στο δικό μου έγγραφο. Δεν πρέπει να τηρήσουμε μόνο το κριτήριο του μήκους, αλλά περισσότερο την ποσότητα των αλλιευμάτων, τον κινητήρα κλπ. Το τζίρο, ε, ατομικές ποσοστώσεις είναι ένα ενδεχόμενο. Επίσης, στη μικρή αλία, όταν θα την έχουμε ορίσει, θα πρέπει να της διαθέσουμε μια ποσόστοση, γιατί μόνο έτσι μπορούν να αξιοποιήσουν τις μπορεί να την αξιοποιήσουν την ποσόστοση. Επίσης, ε, αυτά, αυτά είναι τα πιο βασικά, θα επανέλθουμε. Δεν ανησυχείτε, θα επανέλθουμε στην επόμενη συνεδρίαση. Δεν πειράζει που δεν έχουμε χρόνο τώρα. Ε, Συγχαρητήρια για την έκθεση αυτή, για αυτή την έκθεση εργασία ε, που... Να σας πω ότι δεν είναι κοινή μας γλώσσα, αλλά έχουμε είναι μία από τις κοινέ γλώσσες στην Ιβηρική. Η μικρή παρακτή αλία δεν είναι ίδια γιατί αλλάζει σε διάφορες ε, ζώνες. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη την ε, γεωμορφολογία, τις τεχνικές και τις κοινωνικές πτυχές. Νομίζω ότι ο κ. Φερέιρα αναφέρεται σε αυτή την ε, ε, διαφοροποίηση των κριτηρίων ε, και αναφέρεται σε αυτόν τον ορισμό ο οποίος ε, πρέπει να αλλάξει γιατί είναι επιβαλαιωμένος και θέλω να επιστήσω την προσοχή στο ότι δεν πρέπει να επικεντρώνουμε στη συζήτηση στο τι θα κάνουμε μια εξαίρεση αλλά στο να έχουμε ένα γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Πρέπει να γενικεύσουμε και εκεί πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η μικρή παράκτη ελία e δίνει, δημιουργεί θέσεις εργασίας στο 90% ε, και ε, ξέρετε, εγώ προέρχομαι από την Γαλλική και εδώ δεν ε, συμφωνώ με την κυρία Φράγα γιατί χρησιμοποιούνται εργαλεία επιλεκτικά. Έχει αποδεικτεί αυτό ότι υπάρχουν... Ε, τέτοια επιλεκτικά εργαλεία και αναγνωρίζεται και από το δικό τη ε, κόμμα ότι αυτά τα εργαλεία θεωρούνται επιλεκτικά και δεν το λέω εγώ, το λένε οι οικολόγοι. Ναι. Έτσι λοιπόν πρέπει να αναφερόμαστε και σε αυτό το κριτήριο τη χρήση επιλεκτικών εργαλείων και ιδίω πρέπει να χρησιμοποιηθούν ε, πολιετοί. πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό όταν ε, δημιουργούνται πολιετοί σχέδια για όλα τα αλλιεύματα. Ευχαριστώ κυρία Γκαρσία Γέρο. Τηλεγραφικά. Εξαιρετικό το έγγραφο εργασία κατά την άποψή μου και νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε περισσότερη ευκαιρία και άλλη ευκαιρία να το συζητήσουμε αυτό, ακόμη και άτυπα. Η κυρία Επίτροπος χτες ε, σε καμία περίπτωση δεν αναγνώρισε ε, ότι στην μεταρρύθμιση δεν ε, αντιμετωπίζεται όπως πρέπει το θέμα της ε, μικρής και παράκτητης ελίας. Εμείς συμφωνούμε με τους στόχους σε κοινωνικό επίπεδο, σε οικονομικό επίπεδο και σε ό,τι αφορά την απασχόληση. Αυτή είναι η θεμελιώδης βάση, κυρία βάση και αυτό πρέπει να γίνει και με τη συμμετοχή των ίδιων των αλλιέων, των εργανώσεων των αλλιέων και των οικολόγων. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε και το πώς ε, θα υπάρξει ανανέωση ε, γενολογική, δηλαδή να δώσουμε στους νέους ε, τις ίδιες ευκαιρίες όπως και στους γονείς τους. Και επίση το θέμα των γυναικών, αλλά έχουμε και το Ταμείο της Χρηματοδότησης, πρέπει πραγματικά να συμβάλλει και να βοηθά όσους μπορούν να αναπτύξουν μια βιώσιμη αλία. Ο κ. Αντινόρο. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ δεν θα μπορώ να μπω τώρα σε μεμονωμένα θέματα, δεν έχουμε χρόνο. Γενικά συμφωνώ ε, με το πώς παρουσιάζεται το ζήτημα και τώρα η κυρία Φράγκα είπε ότι είναι δηλιακή εικόνα. Ε, εντάξει, μερικές φορές και μέσω του ονείρου μπορούμε να φτάσουμε στη λύση. Ε, τώρα τι επόμενε συνεδριάσει ε, για αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέλω να παρακαλέσω να έχουμε τον κατάλληλο χρόνο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε όπω πρέπει και να ανταλλάξουμε απόψει, γιατί με αυτόν τον τρόπο σε τίποτα δεν εξυπηρετεί. Δηλαδή μετά παρουσιάζουμε κάποιες τροπολογίες αλλά δεν έχουμε μπορέσει να εργαστούμε πριν. Ευχαριστώ που τηρήσατε και το χρόνο. Κομισιόν, κύριο Κούπερ. Ευχαριστώ. 30 δεύτερα μόνο. Να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική πρωτοβουλία. Η ανάδειξη της σημασίας του στόλου μικρής κλίμακας είναι σημαντικό και για εκείνον και για την Κομισιόν. Το είπαμε πολλές φορές, αναγνωρίζουμε την αξία, την σημασία, τις ιδιαιτερότητες του στόλου μικρής κλίμακας. Εδώ ευθυγραμμιζόμαστε απόλυτα. Ε, πιστεύω ότι η έκθεση έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, πρέπει να τα συζητήσουμε περισσότερο και να φωτίσει και η Κομισιόν, να διαφωτίσει την Κομισιόν και τον εισηγητή ε, δίνοντας απαντήσεις σε κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα ε, που αναφέρονται στην έκθεση Φερέιρα και προσβλέπουμε στη συζήτηση αυτή. Ας σταματήσω καλύτερα εδώ και την επόμενη φορά ελπίζω να έχω περισσότερο χρόνο. Ευχαριστώ. Τέλος, ο κύριος Φεραίρα. Δεν έχω και πολλά να πω. Δυστυχώς δεν είχαμε χρόνο επαρκή. Ελπίζω να έχουμε σε μια άλλη συνεδρίαση λίγο περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε την έκθεση. Αν όχι, θα ήθελα να σε επενθυμίσω, δεν πρόκειται ακόμη για σχέδιο έκθεση, είναι ένα έγγραφο εργασίας και σίγουρα θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες μελλοντικά για να συζητήσουμε. Ούτως ή άλλως είμαι στη διάθεσή σας. Αν έχετε κάποια ε, πιο λεπτομερή θέση, επικρίση, οτιδήποτε θέλετε να μου δώσετε ω υλικό, είμαι στη διάθεσή σας σας Να πω μόνο κάτι. Σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Φράγα για την ιδηλιακή έτσι, αντιμετώπιση του ζητήματος από πλευρά. μου, ήθελα να σας πω, να σας παραπέμψω στο έγγραφο εργασίας, εκεί που λέω ότι, τέλος πάντων, να το πω αλλιώ. παραδέχομαι ότι υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση και ότι υπάρχει, υπάρχουν διάφορα είδη αλίας μικρής κλίμακα. Δεν μπορούμε όλα να τα εξισώνουμε. Λοιπόν, άρα πρέπει να ορίσουμε καλύτερα ποια είναι η μικρή αλία, ποιος ψαρεύει, πού ψαρεύει, πώ ψαρεύει, ποια, ποιες είναι οι περιοχέ όπου όντω μπορεί να χαρακτηριστεί η αλία ως αλία μικρή κλίμακας. Όντω υπάρχει ένα θέμα ορισμού, ένα κενό αν θέλει στην νομοθεσία και πρέπει να το καλύψουμε. Ο κύριος Στίβενσον, ευχαριστώ το ότι συμμετείχαν 10 άτομα στη συζήτηση παρά τον ελάχιστο χρόνο. Ε, καταδεικνύει το ενδιαφέρον τη Επιτροπή. Γι' αυτό το ζήτημα την επόμενη φορά θα τα πούμε. Ευχαριστώ και τι διερμηνεί που μα έδωσαν λίγη περισσότερη ώρα. Ευχαριστούμε και εμεί. Θα ήθελα να σα επενθυμίσω ότι αρχίζουμε και κλεισμένο των θυρών για την συζήτηση που θα γίνει για τι διεθνεί διαπραγματεύσει. Τρει η ώρα και κλεισμένο των θυρών. Το θυμίζω. Ευχαριστώ. Γεια σα.